Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Βάσει της ημερησίας διάταξης προχωρούμε στην κοινή συζήτηση για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Καταστατικό της Ρώμης. Με την έκθεση του κύριου Ραμών Χαουρέγγι, για τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του και των θεμελιωδών ελευθεριών και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την διάσκεψη για την αναθεώρηση του καταστατικού της Ρώμης σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Καμπάλα της Ουγκάντα. Δίδω αμέσως το λόγο στον εισηγητή κύριο Χαουρέγγι για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ κύριε Σίγητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου. Νομίζω ότι η μέρα αυτή είναι μια σημαντική ημέρα. Ξέρω ότι πολλές είναι οι σημαντικές μέρες στο σώμα αυτό. Νομίζω ωστόσο ότι από τη στιγμή που εγκρίθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου, η εντολή για να μπορέσει η Ένωση να ε, προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί ένα από τα μεγάλα νέα της διαδικασίας ενοποίησης της Ευρώπης και οικοδόμησης της Ενωμένης Υπήρου μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι φτάνουμε στην κορύφωση μιας παλιάς προσδοκίας που αποτελεί τμήμα του ιστορικού πυρήνα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Διότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα του ανθρώπου, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν τμήμα του DNA της ευρωπαϊκής ιδέας. Η έκθεση που θα εγκρίνουμε αύριο και που συζητούμε σήμερα έχει στόχο να θεσπίσει την εντολή αυτή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ε, συνθήκη της Λισαβόνης και μετά. Και εγώ θέλω να συνοψίσω το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής με τρεις βασικές ιδέες. Πρώτον, να υπενθυμίσω ότι δεν είναι τα κράτη-μέλη μόνο αυτά που προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νέα νομική της προσωπικότητα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας το κοινοτικό δίκαιο και η ανάπτυξη του κοινοτικού κεκτουμένου που υπόκεινται πλέον στις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάτω από την, τον έλεγχο ενός δικαστηρίου εκτός της Ένωσης που πάντα εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών αυτών. Δεύτερον, την ε, συμβολή την ε, χορήγηση μάλλον στους Ευρωπαίους πολίτες ενός νέου δικαιώματος και ενός νέου ε, δικαστηρίου στο οποίο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για να ζητήσουν την τήρηση των ε, νέων αρχών που περιλαμβάνει η Ένωση έναντι των κρατών ή έναντι της Ένωσης. Τρίτον, το ότι οι δραστηριότητες εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δραστηριότητες αστυνόμευσης και ασφάλειας εκτός των συνόρων μας, και η διεθνή συνεργασία υπόκεινται και αυτέ τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει κατά την άποψή μου, κυρίε και κύριοι, ότι έχουμε κάνει ένα ιστορικό άλμα προ τα εμπρό στην διαδικασία ενοποίηση, στην οικοδόμηση τη ουσιαστικότερη ιδέα τη Ευρώπη που, όπω έλεγα προηγουμένω, απαντά στις απαιτήσει των Ευρωπαίων πολιτών και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεύτερον, απαιτεί μια ενίσχυση, εμπεριέχει μάλλον μια ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι μαζί με το Χάρτη Δικαιωμάτων και την προσχώρηση στη συνθήκη της Λισαβόνας, από κοινού δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο σχεδόν τέλειο και κατά συνέπεια το πλέον προηγμένο πλαίσιο προστασία του κόσμου. Ενισχύοντα την αξιοπιστία τη Ένωση έτσι έναντι τρίτων χωρών, όπου στι διμερεί τη σχέση η Ένωση πάντα απαιτούσε να τηρούνται ε, οι αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η έκθεση αυτή ε, παρουσιάζει περιλαμβάνει μάλλον θεσμικές και νομικές διαστάσεις που δεν θα παρουσιάσω. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ξεκινά πλέον μια διαδικασία. Διότι η Επιτροπή, και ευχαριστώ την κυρία Ρέντινγκ για την ταχύτητα με την οποία ενεκρίθη η εντολή της διαπραγμάτευσης και το Συμβούλιο που θα κάνει σύντομα με την έκθεση αυτή που ξεκίνησε και με την ε, ε, εξωτερική με την, υπηρεσία, με την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και ευχαριστώ τους συζητητές γι' αυτό, μας δίνει ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να έρθει η σύμβαση προσχώρησης γρήγορα στο Κοινοβούλιο ξανά και να προσχωρήσουν και τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός κ. Λόπες Γκαρίντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως έλεγε και ο κύριος Χαουρέγγι, η σημερινή συζήτηση και αυτή που μόλις έγινε θα έλεγα στην Ορομέλεια είναι μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση που αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Όταν δηλαδή θεωρούμε ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι πλέον αρμοδιότητα των κρατών, που είναι ο κύριος πολιτικός ε, παράγοντας των τελευταίων αιώνων, αλλά γίνεται αρμοδιότητα της ανθρωπότητας. Ξεπερνάει τα σύνορα και δημιουργεί μια σειρά θεσμικών εγγυήσεων για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δικαιώματα του ανθρώπου, η ΕΣΒΑ δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αποτελεί έναν από τα πιο πολύτιμα εργαλεία της Ευρώπης και η διεθνής και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι παραδείγματα μεγάλων βημάτων μπρος για την παγκοσμιοποίηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της προστασίας τους. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν έχω να προσθέσω πολλά σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Χαουρέγγι. Δεν θέλω να προσθέσω ιδίω ε, περισσότερα στην εξαιρετική έκθεσή του, τόσο του ιδίου όσο και των άλλων εισηγητών, κύριων Κριστιαν Πρέντα και Κίνγκα Γκάλ, για το ζήτημα αυτό της υπογραφής από πλευράς Ένωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θέλω να επαναλάβω πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Χαουρέγγι. Να υπογραμμίσω ότι η προσχώρηση είναι ένα στοιχείο ενοποίησης, μια ενίσχυση κατά συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιπλέον θα, προσ... θα προστεθεί στην μεγάλη καινοτομία της συνθήκης της Λισαβόνας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που θα αποτελέσει που θα δουλέψουν από κοινού και θα είναι ένα από τα τεχνικά έργα του, της προσχώρησης αυτής, τη δυνατότητα δηλαδή συνεργασίας του Δικαστηρίου της Ένωσης και του ΕΔΑΔ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, χωρίς κάποιος να παραχωρήσει κάτι. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας αυτής οδηγεί σε αύξηση της αξιοπιστίας της Ένωσης στον τομέα της πρόσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μην ξεχνάτε ότι εμείς ζητάμε από τρίτες χώρες της Ευρώπης που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ε, ΕΣΔΑ. Η πρότασή μας εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται. Με την προσχώρησή μας η Ένωση και όχι μόνο τα μέλη της Ένωσης, υπόκειται και αυτή στη δικαιοδοσία του ΕΔΑΔ, του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το υπογραμμίζει πολύ σωστά αυτό ο κ. Χαουρέγγι. Σε ό,τι αφορά το θέμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Βρισκόμαστε πάλι σε ιστορική στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό Γεγονό, σε λίγε μέρε ξεκινά η διάσκεψη αναθεώρηση του καταστατικού τη Ρώμη. Είναι η μόνη διάσκεψη που είναι υποχρεωτική και πρέπει να υιοθετηθεί για την αναθεώρηση του καταστατικού τη Ρώμη και για την επίτευξη μια ισορροπία σε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, την, ε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Βρισκόμαστε λοιπόν, έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα ε, γεγονός τεράστιας σημασίας που εξετάζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο COPS και αύριο θα περάσει στην Κορεπέρ. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί το ψήφισμα από πλευρά Συμβουλίου. Θα συμφωνήσουμε με αυτή την προσέγγιση μην ξεχνάτε ότι πέραν ημών και άλλα κράτη εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, ε, της Λατινικής Αμερικής στα πλαίσια του οργανισμού UNASUR. Μην ξεχνάτε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αντιστοιχεί, ανταποκρίνεται σε μία δέσμευσή μας για ε, τιμωρία των ε, σημαντικών ε, αδικημάτων κατά της ανθρωπότητας από όλους τους ε, από όλες τις χώρες της Ένωσης. Το 2003 το 2004 υπήρχε ένα σχέδιο δράσης και μια συμφωνία συνεργασίας με το δικαστήριο του 2006. Όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης σήμερα αποτελούν συμβαλόμενα μέρη ε, του καταστατικού της Ρώμης και υπόκειται κατά συνέπεια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για να υπογραμμίσουμε το ρόλο που έχει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στον κόσμο και τη δέσμευση της Ένωσης για την ενίσχυση του δικαστήριου αυτού που αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με την Αφρικανική Ήπειρο αλλά η διάσκεψη στην Καμπάλα θέλει να πει στους Αφρικανούς ότι δεν είμαστε κατά της Αφρικής αλλά με την Αφρική. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η διάσκεψη αναθεώρηση του καταστατικού που είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη, την κοινωνία των πολιτών, τους περιφερειακούς οργανισμούς και που επιτρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση της κατάστασης τη διεθνού δικαιοσύνη τη στιγμή που το δικαστήριο αυτό ε, γίνεται το μόνο διεθνέ μόνιμο ποινικό δικαστήριο στον κόσμο. Ε, το μόνο διεθνές ποινικό δικαστήριο στον κόσμο. Ευχαριστώ. Η επίτροπο κυρία Ρέντινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους ομιλητές, με όλους όσους εργάζονται για το θέμα αυτό. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι συνταγματικής σημασίας. Το σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, μέσω της Συμφωνίας της Λισαβόνας, της συνθήκης Λισαβόνας, δεν αφήνει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πλέον υποχρέωση. Είναι λοιπόν πολύ θετικό γεγονός το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή αυτής της διαδικασίας έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται και από το ψήφισμα που έχει υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους εισηγητές της Επιτροπής ε, Ελευθεριών και συνταγματικών υποθέσεων, καθότι οργάνωσαν και μία ακρόαση η οποία ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Αουρέγγι είναι σε μεγάλο βαθμό ένα κείμενο το οποίο συμβαδίζει με τις προτάσεις της Επιτροπής. Υπάρχουν τρία σημεία που κατά την άποψή μου έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, η Επιτροπή συμφωνεί ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στα προσθετικά πρωτόκολλα, τα οποία δεν έχουν κυρωθεί από όλες τις χώρες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Αυτό για την άσκηση της ε, των αρμοδιοτήτων και της εξουσίας των ε, δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που φαίνεται και από την χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε κάποιες διατάξεις έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να προσχωρήσει σε αυτά τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα σε ποια θα προσχωρήσει de facto, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί ομόφωνα από το Συμβούλιο, αφού προηγουμένως δοθεί σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η ιδανικό θα ήταν όλα αυτά τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα να ληφθούν μαζί υπόψη Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτονομία, με δικές της εξουσίες, σαν ένα συμβαλόμενο μέρος, το οποίο αρχικά έχει προγραμματιστεί και σχεδιαστεί για κράτη-μέλη. Κάποιες τεχνικές προσαρμογές, διαδικαστικές αν θέλετε, είναι απαραίτητες όσον αφορά αυτήν την ειδική προσχώρηση και την ειδική νομική φύση του κοινοτικού δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν οι μηχανισμοί, οι αντίστοιχοι μηχανισμοί, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η προσαρμογή και, το η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει με αντιστοιχεία να εφαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι προτάσεις συμβαδίζουν με την πρόταση της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Τρίτον, συμφωνώ απολύτως με αυτό που προτείνει η έκθεση, δηλαδή συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης όρις με όλα τα υπόλοιπα συμβαλόμενα μέρη. Αυτό είναι προϋπόθεση για την ομαλή ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα της σύμβασης. Καταλάβατε οπωσδήποτε πιστεύω ότι η παρουσία ενός δικαστή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκπροσωπεί όλα τα συμβαλόμενα μέρη προϋποθέτει και έναν δικαστή ο οποίος εκλέγεται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ίσα δικαιώματα και ίσο καθεστώς, ίδιο καθεστώς με τους υπόλοιπους δικαστές. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου. Όπως προβλέπει η σύμβαση, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου θα εκλέξει έναν υποψήφιο μετά από τρεις υποβολές υποψηφιότητας από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως θα πρέπει να συμμετάσχουν αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτής της εκλογής. Η εκλογή από έναν κατάλογο τριών υποψηφίων είναι θέμα που θα πρέπει να γίνει με εσωτερικούς κανόνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης, όπως προβλέπει το άρθρο 255, να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξάλλου η διαδικασία για την εκλογή του δικαστή, των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ισπανική Προεδρία θεωρεί το θέμα αυτό ύψη τη προτεραιότητα. Η Ισπανική Προεδρία θα ήθελε να υπάρξει συμφωνία πριν το τέλο Ιουνίου. Εάν το Συμβούλιο μπορέσει να λάβει την απόφαση πριν το τέλος Ιουνίου και το ελπίζω, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση ακριβώς μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπως είπα και πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή σαν διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μας θέματα. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε όμως και το θέμα των διεθνών υποθέσεων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε ότι το 1998 130 χώρες έκαναν ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση υιοθετώντας το καθεστώς που για πρώτη φορά δημιούργησε ένα μόνιμο ποινικό δικαστήριο για άτομα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο άρχισε να λειτουργεί το 2003. Και τώρα έχουμε τη διάσκεψη αναθεώρησης στην Καμπάλα, 7 χρόνια αργότερα δηλαδή, που μας ε, καλεί να κάνουμε μια έγκαιρη ανάλυση των δραστηριοτήτων του δικαστηρίου, των προκλήσεων ε, και την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά τη δράση του δικαστηρίου. Ξέρουμε ότι το δικαστήριο λειτουργεί πλήρως, αλλά βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Και ε, δεν υπάρχει δικαστικός κύκλος που να έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εξετάσει ε, περιπτώσεις πέντε χωρών. Ε, μία δίκη έχει ξεκινήσει, μία άλλη θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και μία άλλη περίπτωση είναι στην προδικαστική φάση. DAR και DRC. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι πρόκειται για ένα δικαστήριο τελευταίας προσφυγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις το δικαστήριο λειτουργεί ως καταλήτης για τις χώρες ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν και να εκδικάσουν υποθέσεις στα εθνικά δικαστήρια. Από την άλλη, στη σύντομη ζωή του το δικαστήριο λειτουργήσε ως φορέας αποτροπής διάπραξης άλλων φοβερών αδικημάτων ε, και ε, με την έννοια αυτή αντιμετωπίζει προκλήσεις. Τώρα, η επικύρωση από πλευράς Μπαγκλαντέζ ε, ανέβασε τον αριθμό των χωρών που έχουν επικυρώσει ε, ε, τη Συμφωνία 111. Ωστόσο απαιτείται η οικουμενική ε, επικύρωση και απαιτείται η συμμετοχή όλων των κρατών μερών, όπως επίσης και όλων των διεθνών φορέων. Το δικαστήριο δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του χωρίς προηγουμένως οι χώρες μέλη να συλλάβουν ας πούμε αυτούς εναντίον των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ούτε αν δεν υπάρχουν ε, φυλακές για να φυλακιστούν αυτοί οι οποίοι καταδικάζονται και γι' αυτό ακριβώς τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ε, προσπαθούν να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει ως βάση, γιατί από την αρχή ήμασταν υποστηρικτές, θεναροί υποστηρικτές της δημιουργίας και λειτουργίας αυτού του Διεθνούς Δικαστηρίου και για να καταπολεμηθεί η ατιμορρησία διότι όπως δείχνει η ιστορία εκατομμύρια άνθρωποι υπέστησαν αυτά τα αδικήματα ελάχιστοι όμως από τους δράστες δικάστηκαν έτσι λοιπόν η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να καταπολεμήσει την ατιμορρησία και να προαγάγει μια διεθνή τάξη βάση του νόμου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υποστηρίζουμε το δικαστήριο, χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα και εργαλεία που διαθέτουμε, ο υπουργό ήδη τα ανέφερε, έχουμε την κοινή θέση που μεθερμινεύθηκε σε ένα πρόγραμμα δράσης. Υπήρξαμε ο πρώτος οργανισμός που που εισήλθε σε συνεργασία και βοήθεια με το δικαστήριο το 2006 και ε, δίδουμε προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πλήρη πολιτική και διπλωματική υποστήριξη με δημοκρατικά διάλογο, με δηλώσεις, με συμπερίληψη των ρητρών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στις διεθνείς συμφωνίες και αυτή πλέον είναι στάνταρ πρακτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το έτος 2000 η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και στη συνέχεια το Μέσο Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα διέθεσε 29 εκατομμύρια ευρώ για έμεση και άμεση βοήθεια ε, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα της κοινωνίας των πολιτών. Ε, Στον τομέα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία ώστε να διερευνηθούν και να ε, δικαστούν να δικαστούν ε, τέτοια ε, αδικήματα. Βεβαίως το σύστημα απαιτεί βελτίωση και δέσμευση από πλευράς όλων των χωρών του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει ο κύριος Πρέντα για την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών για δύο λεπτά θα μιλήσω πρόεδρε για την έκθεση Χαουρέγγι και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση, εξαιρετική έκθεση που με εξαντλητικό τρόπο εξετάζει τα υπέρ και τις προκλήσεις της προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ. Ήμουν εισηγητής προς γνωμοδότηση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω το βασικό πλεονέκτημα της προσχώρησης της Ένωσης στη Σύμβαση. Μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν αυτονόητο. Πρόκειται όμως για μια ελπίδα που επαναλαμβανόταν 30 χρόνια. Ελπίζω ότι η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ θα βελτιώσει το διάλογο της Ένωσης με τις τρίτες χώρες και θα δείχνει σε όλους ότι η Ένωση είναι μια κοινότητα δικαίου τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης θα τα, όργανα της Ένωσης θα ελέγχονται από το δικαστήριο του Στρασβούργου με βάση ενιαίους κανόνες σεβασμού του δικαι... των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η προσχώρηση στην σύμβαση αποτελεί για να, ε, ευκαιρία για να προσχωρήσει η Ένωση και σε άλλα συμπληρωματικά πρωτόκολλα. Την αναφερειμένη κοινωνική χάρτα, για παράδειγμα, που προσφέρει προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον πιστεύω ότι η Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα των οργάνων του Συμβουλίου, να μετάσχει στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και αυτό θα έχει θετική συνέπεια στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όπως αναφέρει και η έκθεσή μου, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του ειδικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και της διαφύλαξης του δικαιοδοτικού συστήματος του Στρασβούργου που έδειξε την αποτελεσματικότητα στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Γκάλ για την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και για δύο λεπτά έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. Πιστεύουμε πραγματικά ότι αν οι δύο επιτροπές μας συνεργαστούν και συνεργαστούμε και με την νομική επιτροπή θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν την προσχώρηση στην σύμβαση και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα ακόμα εκρεμή θέματα. Εγώ σας μιλώ εξ ονόματος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Ελευθεριών και θα ήθελα εδώ να θίξω τα θέματα που για μας είναι τα πιο σημαντικά. Θεωρούμε ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το πολύ σημαντικό και περιέχει πολλά πλέον εκτήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της προσχώρησης και ποιε είναι οι θεμελιώδεις αξίε τις οποίες θέλουμε να προασπιστούμε. Απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει να δώσουμε αβάσιμες ελπίδες. Τι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για το μέλλον. Καταρχήν τις σχέσεις μεταξύ του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του, Λουξεμβούργου και του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Καθότι δεν πρόκειται να να αλλάξει η δικαιοδοσία των δύο αυτών δικαστηρίων στο μέλλον. Θα μεταρρυθμιστούν τα δύο αυτά δικαστήρια κατά τη διάρκεια της προσχώρησής μας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα είναι χρήσιμο για όλους εάν βεβαίως όλοι οι θεσμοί κάνουν αυτό που πρέπει. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση είναι κάτι το μοναδικό. Είναι όμως κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητήσει όλα αυτά που έχουμε κάνει ήδη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ό,τι γίνει από εδώ και πέρα θα πρέπει να θεμελιώσει και να ενισχύσει αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν και επαναλαμβάνω είναι μια προστιθέμενη αξία σε αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μπαίνουμε τώρα στους αγωγητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ξεκινά η κυρία Ένε. Δύο λεπτά για το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πέτροπε, το η αναθεωρητική διάσκεψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι ιδιαίτερη σημασία για... και για το δικαστήριο αλλά και ε, για την ε, διεθνή ε, κατάσταση. Θα επανεξετάσει το έργο και τις δραστηριότητες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και θα προτείνει λύσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Καταρχήν η συμμετοχή των διατλαντικών μας εταίρων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα αν έχει τη δική τους υποστήριξη. Θα πρέπει λοιπόν οι Αμερικανοί εταίροι μας να ξεκαθαρίσουν τη δική τους εμπλοκή στο ε, ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ. Επίσης, θα πρέπει να δούμε το άρθρο 104 με βάση το καταστατικό της ε, Ρώμης που επιτρέπει στις χώρες μέλη να ε, λάβουν μέτρα με βάση την ε, νομολογία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί από το καταστατικό της Ρώμης. Και τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή του καταστατικού της Ρώμης και την ενσωμάτωση στην νομοθεσία των χωρών που δεν το έχουν πράξει ακόμα, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ε, κατά τη διαδικασία διεύρυνσης ε, της ε, ε, Ένωση. Η ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην Ρωσία, διότι αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε τους ε, τρόπους της εταιρική σχέσης με τους Ρώσου εταίρου μα. Ευχαριστώ πολύ. Για την Συμμαχία Προοδευτικών Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Σερακιάνη, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την προσχώρηση τη Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αποτελεί ένα υπέρ για του Ευρωπαίου πολίτε, γιατί χάρη σε αυτό θα έχουν ένα νέο δικαστήριο έξω τη εκτός Ένωση που θα εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα των πολιτών τη Ένωση θα, γίνονται σεβαστά από την Ένωση και τα κράτη-μέλη. Βάσει των αρχών τη Δημοκρατία, η Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν πάντα το δικαίωμα να υπερασπίζονται αυτού. Γι' αυτό είναι θεμελιώδε Κάθε κράτος που προσχωρεί στη συνέλευση, στην σύμβαση να έχει και ένα δικό, δικό του ε, δικαστή. Γι' αυτό είναι σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ένα άτυπο όργανο για να, για να συντονίζει τι συζητήσει μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Επιπλέον είναι σημαντικό να εμπλακεί το Κοινοβούλιο στι διαπραγματευτικέ διαδικασίε. Να προσθέσω επιπλέον ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν το δικαίωμα να, να καταλαβαίνουν Τέτοιου μηχανισμού και το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό θεωρώ θεματικό, το, σημαντικό το Συμβούλιο της Ευρώπης και Ένωση να εξετάσουν το δεχόμενο να διαμορφώσουν κατευθείαν γραμμέ που θα εξηγούν σε όλους ότι τις συνέπειες μιας τέτοιας προσχώρηση. ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους και δημοκρατικούς, ο κύριος Ντάφ, 1,5 λεπτό η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, ΕΣΔΑ αναμένεται το μακρόν. Πρόκειται για ε, ένα σημαντικό ε, βήμα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επίσης ε, με την εξωτερική εποπτεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα. διότι θα καταστήσει δεσμευτικό το περιεχόμενο της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα δώσει νέα πνοή. Ε, στην ε, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό το υποστηρίζουμε εμείς οι Βρετανοί φεντεραλιστές οι οποίοι είμαστε υπέρ της υπερεθνικής προσέγγισης. Ένας τέτοιος συνδυασμός είναι απολύτως ορθός αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή της πολιτικής της, ε, των συμμαχιών μεταξύ Βρετανών φιλελευθέρων δημοκρατών και συντηρητικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους και ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία, η κυρία Λόχμπιλε, για δύο λεπτά. Όσον αφορά το καθεστώς και την κατεύθυνση του νέου ποινικού δικαστηρίου, μπορούμε να δώσουμε πολλά παραδείγματα. Αυτό όμως που είναι καθοριστικό είναι το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των κρατών, οι εκπρόσωποι της πολιτικής και της στρατιωτικής εξουσίας αποφάσισαν και έκαναν το πρώτο βήμα έτσι ώστε οι εγκληματίες πολέμου και αυτοί που διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας να πρέπει και να μπορούν να προσαχθούν σε αυτό το νέο δικαιωτικό όργανο και στο μέλλον θα πρέπει να συνεχίσουμε την στήριξή μας, να ενισχύσουμε αυτό το νέο δικαστήριο, να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία του. Στην Καμπάλα η συνδιάσκεψη που οργανώνεται θα πρέπει να κάνει μια αποτίμηση αυτών που έχουν πετύχει και αυτών που θα πρέπει να βελτιωθούν. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα κράτη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουν να ομαλοποιήσουν τις διαδικασίες, να θεσπίσουν νέες διατάξεις έτσι ώστε να διευκολύνουν την προσαγωγή των εγκληματιών σε αυτό το δικαστήριο. Επίσης θα πρέπει οι εντολές, τα εντάλματα σύλληψης και όλες οι διαδικασίες να εξομαλυνθούν και να εναρμονιστούν. Το νέο αυτό διεθνές δικαστήριο χρειάζεται συγκεκριμένη στήριξη για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό και να λειτουργήσει η συνδιάσκεψη στην Καμπάλα θα πρέπει να επιληφθεί διαφόρων σημείων όπως ορισμοί των εγκληματών πολέμου και των αρμοδιοτήτων αυτού του δικαστηρίου. Θα πρέπει επίσης να υποβάλουμε ένα κείμενο το οποίο θα περιέχει πολλά από τα σημεία που βρίσκονται σήμερα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί όλους αυτούς τους ορισμού, ορισμούς οι οποίοι θα στηρίξουν την εργασία αυτού του ποινικού δικαστηρίου. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει περιορισμός της ανεξαρτησίας αυτού του δικαστηρίου και θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπροσωπηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο σε αυτήν τη συνειδιάσκεψη. Αυτό θα είναι ένα θετικό μήνυμα και για άλλες περιοχές, αλλά θα δείξει και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Για τους συντηρητικούς και μεθαρισμιστές, ο κύριος Φόξ. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου δεσμεύεται να προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν είμαστε πεπισμένοι ότι, με την, ότι η υπογραφή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσχώρηση στη Σύμφαση είναι ε, ορθό. Ε, εφόσον όλες οι χώρες έχουν συνυπογράψει, τι νόημα έχει να συνυπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήμουν ευχαριστημένος αν κάποιο στην αίθουσα αυτή μου δώσει κάποιο πρακτικό ε, παράδειγμα, αν θα προστατευτούν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα των ε, συμπολιτών μου στην εκλογική μου περιφέρεια, αν υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύμβαση αυτή. Ε, αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωμένες οι χώρες μέλη να ενσωματώσουν την νομοθεσία στην ε, εθνική νομοθεσία. Ε, είμαι βέβαιος ότι αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει αν προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα το Ευρωπαϊκό το, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να υπονομευθεί ο τρόπος με τον οποίο το Βρετανικό Κοινοβούλιο προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα απλώς είναι μια κίνηση για να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ε, πρωταγωνιστής ε, στην διεθνή σκηνή. Κατά τη γνώμη μου όμως αυτό είναι ένας λόγος για να μην υπογραφεί η σύμβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, Πράσινη Σκανδαλική Αριστερά, ο κύριος Σόλτ. Για ένα λεπτό, για ένα μισή λεπτό, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μου ομάδα στηρίζει χωρίς κανέναν ενδιασμό την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για την κοινωνική, για την ανθρωπιστική διάσταση και συμφωνώ απολύτως με τον ε, συνάδελφο τον κύριο Φόξ, ο οποίος λέει ότι κάθε χρόνο χιλιάδες προσφυγές επιβαρύνουν το δικαστήριο του Στρασβούργου και ότι οι αποφάσεις καθυστερούν λόγω φόρτου εργασίας. Ακριβώς αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, το οποίο όμως δεν είναι αρμόδιο για θέματα θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το δικαστήριο του Λουξεμβούργου σε καμία περίπτωση δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο παρελθόν για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς ε, θα πρέπει εδώ να χαρακτηρίσουμε αυτή την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν ιστορικό γεγονός και ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτήν την προσχώρηση καθότι με το δικαστήριο αυτό συνεργάζονται και συμμετέχουν οι χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, συν όλες οι χώρες οι οποίες συνεργάζονται στα πλαίσια της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αυτού του νέου δικαστηρίου και οι διαδικασίες θα πρέπει να βοηθήσουν έτσι ώστε με σύντομο και επικοδομητικό τρόπο να βρεθούν λύσεις στα περίπλοκα τεχνικά και νομικά θέματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Για την Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, ο κύριος Μέσες Μιτ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σίγουρα ε, υπάρχουν υπέρ στην προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση. Αν, για παράδειγμα, απολυθούν οι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ε, κάτι έκαναν. Χάρη στο άρθρο 6 μπορούν να, να προσφύγουν. Άλλοι μπορεί να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν ε, τεράστια πρόστιμα. Αυτοί όμως δεν μπορούν να επικαλεστούν το άρθρο 10 εγώ ωστόσο δεν υποστηρίζω την προσχώρηση της Ένωσης ε, στην σύμβαση γιατί τα κατά είναι πολύ περισσότερα από τα υπέρ. Σίγουρα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ε, το, η προσχώρηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ένας ως ένα, ως ένα επιχείρημα για να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει τα δικαιώματα των πολιτών να μην ε, ενταχθούν σε ευρωπαϊκές ευθύνες. Αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σινκλέρ για τους μη γεγραμμένους. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εισηγητής ανθέσει στην έκθεσή του ότι η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ θα ενισχύσει τους πολίτες κατά των δράσεων της Ένωσης. Εγώ θα ήθελα να προστατεύσω τους πολίτες της δικής μου εκλογικής περιφέρειας από τις δράσεις της ΕΣΔΑ. Στη Βρετανία βεβαίως έχουμε ενσωματώσει το 98 την ΕΣΔΑ που ισχύει σε όλα τα δικαστήρια. Στο... Η νέα κυβέρνηση των συντηρητικών είχε προτείνει να δημιουργήσει ένα νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όπως διαπιστώθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερες ε, ε, αρμοδιότητες στην Βρετανία. Όπως λέει και ο Όργουελ, κάποιοι είναι πιο ίσοι από άλλους σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο ξεκίνημα του μήνα, ε, στην εκλογική μου περιφέρεια, ορισμένοι ταξιδιώτες όπως τους λένε, περιπλανόμενοι δηλαδή, μπήκαν στο, στα σπίτια, στο σπίτι ενός ε, πολίτη της περιοχής μου, αλλά οι άνθρωποι αυτοί, χάρη στην ΕΣΔΑ, έχουν ειδικά, ειδικά προστατευμένα δικαιώματα ε, ε, ε, εις βάρος των φορολογούμενων. Θα έπρεπε αναφέρεται ο εισηγητής στην εμπλοκή των εθνικών διοικήσεων των στην διαδικασία αυτή. Μήπως θέλει να έρθει στην εκλογική μου περιφέρεια ο, ο εισηγητής και να δει πώς οι άνθρωποι αυτοί ε, ε, παραβιάζουν την ιδιοκτησία των συμπολιτών μου. Να δει την αστυνομία που χρησιμοποιείται για να διαφυλάξει την ειρήνη και να προφυλάξει βεβαίως τα δικαιώματα των περιπλανόμενων. Να εξετάσει το πώς οι δρόμοι ε, ερημώνονται να περνούν αυτοί οι άνθρωποι και να προεξοφλώντας τις ε, εγκληματικές δραστηριότητε που έχουν ε, που εμφανίζονται στην περίπτωση που εμφανίζονται αυτοί οι περιπλανόμενοι. Ας εξετάσουμε όταν συζητούμε το θέμα των ειδικών δικαιωμάτων μιας ομάδας πολιτών σημαίνει αυτόματα ότι μειώνουμε τα δικαιώματα των υπολείπων. Δεν θα έπρεπε μία αιρετή εκπρόσωποι να αποφασίζουν ποιο έχει ειδικά δικαιώματα και ποιο όχι. Έχουμε στην Βρετανία μια νέα κυβέρνηση που έδωσε μια σειρά υποσχέσεων. Στο όνομα τη δημοκρατία α υλοποιήσουν τι υποσχέσει του. Ευχαριστώ. Grazie, diamo ora la parola agli altri ε, ε, Παρακαλώ να σέβεστε το λόγο ομιλίας, ε, το χρόνο ομιλίας που έχετε. Για δύο λεπτά ο κύριος Μέντες Δεβίγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν 23 χρόνια είχα την τύχη να μετάσχω στο άλλο κτίριο, στην υπογραφή μια συμφωνία του τότε Πρόεδρου της Επιτροπής κύριου Ντελόρ και του Μαρθελίνο Ρέχα, Γενικού Γραμματέα του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης για την προσχώρηση τότε της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τότε είχε απαντήσει ο κύριος Χάινε όταν τον ε, είχαν ρωτήσει πού θέλετε να πεθάνετε και απάντησε στην Αγγλία, διότι όλα γίνονται με 11 χρόνια καθυστέρησης. 200 χρόνια καθυστέρησης ήταν κάποιες παρεμβάσεις όπως αυτή που ακούσαμε προηγουμένως. Κυρία Πρόεδρε, η ομάδα μου, η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο είναι υπέρ τη προσχώρηση αυτή, Καθυστέρησε πολύ. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έκθεση Χαουράγκη. Ελπίζω να, είναι, να μην είναι τελευταία. Και την καλωσορίζουμε διότι αυξάνει τι εγγύησει των πολιτών. Διότι μπαίνει σε, περισσότερες, σε περισσότερα δικαιώματα στου πολίτε, ώστε η ε, νομοθεσία της Ένωσης να ε, τηρεί τον πίνακα δικαιωμάτων, αυτό τον κατάλογο δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΕΣΔΑ. Η έκθεση ανοίγει το δρόμο για την επίλυση πολλών από τα προβλήματα τεχνικού και νομικού χαρακτήρα που θα εμφανιστούν. Μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση έχει, ε, έχει διαμορφωθεί σε σύμβαση μεταξύ κρατών μελών. Οι κουβέντες που ακούγονται εδώ δεν αφορούν Παρότι αυτά, παρόλο μάλλον αυτά που ακούγονται συχνά εδώ ότι η Ευρώπη είναι ένα υπερκράτος, δεν συμβαίνει. Δεν, δεν ε, ισχύει. Θα σας μιλήσουμε συγκεκριμένα, θα τα πει και η κυρία Γιαννάκου που είναι αρμοδιότητα, το ίδιο είπε και η κυρία Ρέντινγκ για το Συμβούλιο. Χρειάζεται να δοθεί εντολή στην Επιτροπή γρήγορα, ούτω ώστε να προχωρήσει γρήγορα η προσχώρηση της Ένωση της σύμβαση. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιγιάρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους συγχαίροντας τον κύριο Χάουρη και τους συνεισηγητές. Θεωρώ επίσης και εγώ ότι όπως ασχοληθήκαμε με την οικονομική κρίση και την νομισματική κρίση στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να πούμε η Ευρώπη δεν είναι το νόμισμα, δεν είναι η οικονομία, είναι οι πολίτες. Το κείμενο που συζητούμε εμείς ενισχύει την ηθαγένεια. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ένας Bill of Rights για τα δικαιώματα των πολιτών. Ενισχύεται με την εντολή που δίδει το άρθρο 6 της συνθήκης να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων της, ε, του ανθρώπου. Η προσχώρηση αυτή δεν μειώνει κανένα από τα θεμέλια δικαιώματα που εξασφαλίζουν τα κράτη-μέλη στους πολίτες από το γεγονός του ότι είναι πολίτες των κρατών μελών. Αντίθετα, πολλαπλασιάσει και ενισχύει τα δικαιώματα που έχουμε όλοι μας ως μέλη, ως συμμετέχοντες σε ένα κοινό εγχείρημα. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, ως πρόεδρος της, μπορώ να πω ω πρόεδρο τη επιτροπή ΛΥΜΠΟ, ότι ασχοληθήκαμε με όλα τα ζητήματα πλαισίωση τη ΕΣΔΑ στην κοινή αυτή κουλτούρα ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων του πολίτη. Ε, επισκεφθήκαμε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΔΑΔ, επισκέψεις που ήταν εξαιρετικά καρποφόρες. Οργανώσαμε μια τρίτη συνάντηση για 21 Ιουνίου που θα μετάσχουν πολλοί ειδικοί για να έχουμε μια κοινή απόφαση του τι πρέπει να είναι δικαστική προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη. Ένας Βρετανός νομικός, ο κύριος Χάρτ, έγραψε ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς δικαστική εγγύηση. Δεν υπάρχει δικαστική εγγύηση χωρίς δικαστές, όπως δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς πολίτες και δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες αν δεν είναι, έχουν επίγνωση ότι η ευρωπαϊκή οικονόμη, η οικοδόμηση θα υπάρξει μόνο με την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουμε ως μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ενοποίησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάκε για 1,5 λεπτό. λεπτό. Η κυρία Σάκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθώς ε, εξετάζουμε Καθώς μάλλον εξετάζουμε την αναθεώρηση του καταστατικού ε, της Ρώμης, ας δούμε την αποτελεσματικότητα για την ε, δημοκρατία και με την ε, έγκριση από όλες τις χώρες μέλη του καταστατικού θα πρέπει να θέσουμε μπροστά μας και να αξιολογήσουμε το έργο μας ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όμως είναι ένα πολύ σημαντικός φορέας για να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ε, οικουμενικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν την αφοσίωσή του προς την ε, Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, υιοθετώντα κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Είναι πρωταρχική σημασία ε, να ε, διαρευνηθούν και να ασκηθεί δίωξη εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν οργανώσει γενοκτονίε και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προαγάγουμε την προσχώρηση στο καταστατικό ε, ε, της Ρώμης και χώρες εκείνες όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες όπως η Τουρκία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εμπλακούμε σε έναν διάλογο για την ε, παγκόσμια δικαιοσύνη. Ως Ολλανδή θα ήθελα να διαβεβαιώσω τις πολίτες μας ότι ποτέ δεν θα ανακληθεί το ε, έργο του δικαστηρίου της Χάγης. Οι εκτελέσεις, ε, οι βιασμοί και οι ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, γίνονται καθημερινά σε πολλές περιοχές του κόσμου. Θέλουμε λοιπόν η κομμενοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένας σημαντικός φορέας γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν παγκοσμίω να υπάρχει υποστήριξη γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, συνεργάζεται επικοδομητικά για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ πολύ. Να τηρείτε, το, το χρόνο, παρακαλώ, διαφορετικά δεν θα υπάρχει χρόνος για ελεύθερες παρεμβάσεις. Και τώρα το λόγο ο κύριος Άστερ, για να Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ μιλάμε για το δίκαιο και την ομοθεσία σε υπερεθνικό επίπεδο. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρόμοιες περιπτώσεις μου θυμίζουν αυτό που συνέβη στην ίδια μου τη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συνέβη στη Γερμανία, όπου τερατώδη ανθρώπινα όντα στράφηκαν κατά διαφόρων άλλων συμπολιτών τους και πολιτών άλλων χωρών, είτε επειδή ήταν Εβραίοι, είτε επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι, είτε επειδή ήταν φιλελεύθεροι. Και κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφευχθεί, καθότι δεν πρέπει να αφήσουμε κενά στο νομικό μας σύστημα, στο σύστημα της Ευρώπης και θα πρέπει όλοι να ξέρουν ότι υπάρχει ένας δικαστής ο οποίος ξεπερνάει την εθνική δικαιοδοσία και την εθνική νομοθεσία. Αυτό είναι μια τεράστια πρόοδος. Εξίσου σημαντική με την προσχώρηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο πραγματικά εγώ το πολεμάω και το προσπαθώ εδώ και χρόνια. Δεν έχω άλλο χρόνο ομιλία, αλλά ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και ιδιαίτερα τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, το εθνικό μου κόμμα, η συντηρητική, για όσους δεν γνωρίζουν ναι, είμαι συντηρητικός, έχει διατυπώσει σημαντικές επιφυλάξεις για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την δικαιοδοσία του και με βάση το καταστατικό της Ρώμης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες. Ωστόσο, η δέκατη επέτειος μας προσφέρει μια ευκαιρία για να κάνουμε μια σαφή αξιολόγηση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαστηρίου και πράγματι ε, στάθηκε στο ύψος του με διώξεις και με επιδίωξη να συλλάβει τους φοβερότερους τυράννους. Πράγματι ε, βοηθήθηκε το δικαστήριο να λειτουργήσει με αμεροληψία και οι διώξει που ασκήθηκαν υλοποιήθηκαν, κάτι το οποίο βεβαίως ανησυχεί τους Αμερικανούς ε, συμμάχους μας. Ίσως η πρόσφατη σύσταση της ε, συμμαχίας μεταξύ συντηρητικών και φιλελευθέρων μας προσφέρει τώρα μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε τις σχέσεις της Βρετανίας με, την, ε, το Διεθνές Ποινικό ε, Δικαστήριο και στην Καμπάλα να εξετάσουμε αμφίσιμα θέματα όπως είναι η ε, συνυπευθυνότητα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπό ορισμένε συνθήκε το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να διαδραματίσει επικοδομητικό ε, ρόλο σε, στην αποφυγή ενό κλίματο ατιμορρησία για αυτού που διαπράττουν ε, γενοκτονίε ή άλλα ε, αδικήματα κατά τη ανθρωπότητα. Ο κύριος Βερζιά, 1,5 λεπτό. Η κυρία ο 15 λεπτο συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μιλήσω για την ε, προσχώρηση στην, ΕΔΑ, στην ΕΣΔΑ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ποιότητα της ε, δουλειάς που έκανε και τη βούλησή του να ενσωματώσει τις ε, απόψεις των ΜΕΝ και των ΔΕ με συνενετικό πνεύμα. Πέραν των όσων ήδη αναφέρθηκαν για την προσχώρηση, θέλω να υπογραμμίσω δύο σημαντικά για μένα πράγματα. Πρώτον, την ύπαρξη ενός εξωτερικού ελέγχου για την Ένωση και τον εξοδαφικό χαρακτήρα της Σύμβασης, την εφαρμογή της δηλαδή σε όλες τις πράξεις της Ένωσης και εκτός ε, του, του, του, χώρου του, του εδάφους της Ένωσης. Ίσως η δημοκρατία να ενισχυθεί έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η εντολή διαπραγμάτευσης επιτροπής να μην αφορά μόνο τη σύμβαση αλλά και όλα τα πρωτόκολλα ε, της ε, σύμβασης. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ξεκινήσουμε γρήγορα την προσχωρή σε όλα τα νομικά εργαλεία της ε, ΕΣΔΑ για να υπάρχει ένα πλήρες σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δύο ευχές. Πρώτον, η Ένωση να επαγρυπνεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων και των ε, νομικών εκπροσώπων τους. Αυτή, αυτό απαιτεί μια ad hoc ε, νομική συνδρομή με ειδικού ε, ειδικευμένους δικηγόρους. Επιπλέον, η Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε όλα τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν το, την ομοθεσία του στην διεθνή δικαιοσύνη, κάτι που δεν έκανε ακόμα η Γαλλία. Κάτι με λυπεί αυτό, όπω με λυπεί το γεγονό ότι μεγάλα κράτη όπω οι ΗΠΑ δεν μετέχουν στην υλοποίηση τη διεθνού δικαιοσύνη ε, στον τομέα των εγκλημάτων κατά τη ανθρωπότητα. Ευχαριστώ κύριος Μπρόνς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνυπογράφοντας τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα ε, καταστήσει, θα καταστήσει τη Σύμβαση μέρος της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τούτο σημαίνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο θα έχει τη δικαιοδοσία να ερμηνεύσει και να θέσει ισχύ δύο ανταγωνιστικά ε, μεταξύ τους ε, κείμενα, δηλαδή τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον, ε, τη σύμβαση. Έχω ρωτήσει αρκετούς εμπειρογνώμονες ποιο έγγραφο ή ποιο τμήμα θα έχει πρωτοκαθεδρία σε σχέση με το άλλο. Ε, και ε, η απάντηση είναι αυτό το οποίο χορηγεί μεγαλύτερη ευελευθερία. Αργότερα ρώτησα αν έχουμε δύο ε, εταίρους, δύο μέρη σε μια διαδικασία και ας πούμε έρχονται σε σύγκρουση η ελευθερία της θρησκείας και η ελευθερία της έκφρασης. Είναι θεωρητικό βέβαια όπως ε, η περίπτωση ήταν σκίτσων ε, στην Δανία. Ε, και πάλι σε αυτή την περίπτωση η απάντηση ήταν η σιωπή. Είναι σαφές για όλους. Η ελευθερία του λόγου θα θυσιάζεται πάντοτε. Η άρνηση όμως της ελευθερίας του λόγου είναι αυτό το οποίο κάνει καλύτερη η Ευρωπαϊκή Ένωση το πολιτικό δικαίωμα ελευθερίας του λόγου κατά της δίωξης από το κράτος και το δικαίωμα να μην προσβάλλεται κανείς θεωρείται πιο σημαντικό από ότι το δικαίωμα ε, προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Ασκείται βεβαίως ε, κριτική και αυτή η κριτική θα πρέπει να ισχύει και για το ποινικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Γιαννάκου. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο κύριο Ραμόν Χαουρεγγί για την έκθεσή του καθώς και για την καλή συνεργασία που υπήρξε και βεβαίως τους συναδέλφους Πρέντα και Γκάλ για τη συμβολή τους από δύο διαφορετικές επιτροπές. κυρία Πρόεδρε, η ένταξη στην ουσία της ευρωπαϊκής ένωσης στην ευρωπαϊκή συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άρα και στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου απορρέει βεβαίως και από το γεγονός ότι η ένωση απέκτησε ενιαία νομική προσωπικότητα από τη συνθήκη της λισαβόνας. και βέβαια ορισμένοι διαρωτώνται γιατί ενώ ενσωματώσαμε το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων είχαμε ανάγκη να προσχωρήσουμε στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του στρασβούργου καταρχήν το δικαστήριο του στρασβούργου ε, υπό την έννοια του δεδικασμένου έχει αποκτήσει πολύ ευρύτερες δυνατότητες από αυτές που προβλέπονται στα θεμελιώδη δικαιώματα και ήδη το υπενήχθηκαν αυτό τόσο η προεδρία όσο και η επίτροπος κυρία ρέντινγκ. δεύτερον αυτό δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο μια σύνδεση της ίδιας της ευρωπαϊκής ένωσης με τα τεκτενόμενα στο σύνολο της ευρώπης άρα και με τις χώρες που βρίσκονται στο συμβούλιο της ευρώπης. βεβαίως ορισμένοι διαρωτώνται αν αυτό θα δημιουργήσει εμπλοκές γενικότερες αλλά η έκθεση τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν διακρατικές προσφυγές. ούτε τα δικαστήρια είναι το ένα υποκείμενο του άλλου και το άλλο υπερκείμενο το κάθε δικαστήριο έχει αρμοδιότητα στις εξουσίες τις οποίες έχει και άρα και η ευρωπαϊκή ένωση με το δικαστήριο του λουξεμβούργου. θεωρώ ότι είναι ένα ουσιαστικό βήμα αυτό που γίνεται με την προσχώρηση ε, στην δικαιοδοσία της ευρωπαϊκής συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και η διαδικασία για την προσχώρηση στα πρωτόκολλα που αφορούν στις αντίστοιχες εξουσίες και αυτό δίνει τη δυνατότητα βέβαια και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να αναμειχθεί ενεργά στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης καθώς και να συμβάλει μέσω της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του συμβουλίου της ευρώπης στην επιλογή ενός δικαστού. ευχαριστώ πολύ κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χάουιτ για μισή λεπτό. Ε, είμαι επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, για την αναθεώρηση του Διεθνούς Δικαστήριου και ε, αυτό με στόχο την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της ε, ανθρωπότητας και δείχνουμε την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της οικουμενικής δικαιοδοσίας του δικαστήριου. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι 15 από τις 25 χώρες είναι δικές μας χώρες μέλη. Αλλά ταπεινά πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες μέλη που δεν έχουν χρηματοδοτήσει και ούτε έχουν ορίσει ε, ε, εθνικό σημείο επαφής ε, όπως προβλέπει ο χάρτης. Η οικουμενική δικαιοδοσία ξεκινάει από την εφαρμογή εδώ στην ε, Ένωσή μας. Ε, Ένα από, τους, ε, από τα πρώτα θέματα ε, που πρέπει να αντιμετωπίσει η Νέα Βρετανική κυβέρνηση συμμαχίας θα πρέπει να είναι να συνυπογράψει ούτως ώστε να αποτρέψει τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής κατά της ανθρωπότητας Ξέρουμε ότι οι δράστες των ε, εγκλημάτων του Δευτέρου ε, Παγκοσμίου Πολέμου ε, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν από το δικαστήριο της Νερεμβέρχης. Η χρήση ε, δεν ξέρω ε, πώς είναι δυνατόν να καταδικάζουμε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, παράνομα σφαίρες ενώ αυτές επιτρέπονται εντός της επικράτειας. Δράσαμε εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν ενώ από την άλλη οι δράστες μπορούν να λειτουργήσουν ελεύθερα εντός της επικράτειάς μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, έχοντας συσταθεί για να κρίνει και να καταδικάσει τους υπευθύνους διάπραξης γενοκτονιών, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συνιστά μια πρώτη απάντηση προς τα θύματα που απαιτούν ε, και συχνά από κατάσταση και δικαιοσύνη. Υπήρξαμε πολλοί άριθμοι ε, ε, εκείνοι οι οποίοι ζητούσαν έναν προληπτικό ρόλο για το Διεθνές Δικαστήριο πριν από τη δημιουργία του. Πράγματι, ε, ένα δικαστήριο το οποίο θα είχε τη δικαιοδοσία να ε, ασκήσει διώξεις εναντίον ε, φοβερών ε, δραστών εγκλημάτων στη Βοσνία, τη Ρουάντα, την Καμπότζη ή το Νταρφούρ. Δεν θα ήταν και ένας τρόπος για την πρόληψη και παρεμπόδιση επανάληψης τέτοιων αδικημάτων στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν λειτουργήσε αυτή η, αν λειτουργήσε προληπτικό στο δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας γνωρίσει παραδείγματο χάρη αν το ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον του Πρόεδρου Ομάρελ Μπεσίρ συνιστά ένα μέρος της λύσης ή μέρος του τους. Και επίση μπορεί να μας δώσει ε, μια απάντηση για το αν προτίθεται να κάνει τροποποιήσεις στη διάσκεψη στην Καβάλα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριο Πρόεδρε, η προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ πρέπει να αποφύγει μια σειρά κινδύνων που θα προκύψει ενδεχόμενα από τον ανταγωνισμό μεταξύ του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου ή την, ε, τις συγκρούσεις μεταξύ της συνύπαρξης δύο κειμένων της ΕΣΔΑ και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων Ίσως λοιπόν να προκύψουν προβλήματα δικαιοδοτικά και νομικής βάσης. Η προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση θα πρέπει να γίνει με σεβασμό των συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών που θέτουν τους γενικούς κανόνες δικαίου. Η προσχώρηση δε δεν θα πρέπει να καταστρατηγεί το δεσμευτικό πρωτόκολλο της συνθήκης της Λισαβόνας για την ειδική αντιμετώπιση της, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζέγγεντη, Ένα λεπτό. Λυπούμε πάρα πολύ, γιατί έχω μόνο ένα λεπτό για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Παρ' όλα αυτά θα μπορέσω να ασχοληθώ με δύο πολύ σημαντικά σημεία. Θα ήθελα καταρχήν να σας ενημερώσω όσον αφορά τις πλημμύρες οι οποίες πλήττουν την Ουγγαρία και την Πολωνία. Χιλιάδες άτομα απειλούνται. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και εδώ στο Στρασβούργο. Θα πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί και να ζητήσω σε όλους τους υπεύθυνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προτείνουν την υποστήριξή τους και τη βοήθειά τους στα θύματα. Έχουμε 12 πόλεις στο βόρειο τμήμα της Ουγγαρίας που έχουν πληγεί από αυτές τις πλημμύρες, από αυτές τις θεομηνίες και ελπίζω πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να συνδράμει αυτά τα μέρη της χώρας μας. Όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την προστασία του σε πολύ ψηλό επίπεδο, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπινα δικαιώματα, απλώς ενστερνιζόμαστε τα ιδεώδη και τις θεμελιώδεις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ θετικό. Είμαστε αντίθετοι με αυτά τα ιδεώδη και πραγματικά θα πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καζίνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύον του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, βεβαίως η προσχώρηση αυτή είναι μήνα, μήνυμα μιας, ε, του πεπρωμένου της Ένωσης να προασπίσει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πεπρωμένο που περιλαμβάνει η ολόκληρη δομή της και ανατρέχει στην ιστορία της από την εποχή της προσχώρησης των κρατών μελών στην ε, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και την επανειλημμένη αναφορά του ότι οι γενικές αρχές της σύμβασης και που είναι και στα συντάγματα των κρατών μελών αποτελούν πλέον τμήμα του ευρωπαϊκού δικαίου. Η συμβολική αυτή χειρονομία λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Το να μεταφράσουμε όμως σε νομικό κείμενο, συγκεκριμένο νομικό κείμενο, αυτή την πραγματικότητα δεν είναι απλό. Η έκθεση ασχολείται κυρίως και μόνο με τις θεσμικές διαστάσεις της προσχώρησης. Αποδεκτές και σημαντικές. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Χαουρέγγι και πρέπει να τονίσω ότι η Επιτροπή Συνταγματικών υποθέσεων τις οποίες προεδρεύω ενέκρινε ομόφωνα το κείμενο. Μας ικανοποιεί λοιπόν το κείμενο αυτό και δεν θα σταθώ στις επιμέρους διαστάσεις του διότι συμφωνούμε σχεδόν όλα όσα ανέφερε ε, η Επίτροπος και ο Προεδρεύων. Μία πρόταση μόνο. Επειδή έμεινε κάπως ασαφής η δήλωση για την θεσμική παρουσία ευρωβουλευτών στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν, εξετάζει, όταν συναντιέται για την εκλογή των δικαστών. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την σχέση, το συσχετισμό μεταξύ πληθυσμού της Ένωσης και πληθυσμού των υπολείπων χωρών μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Βεβαίως, η παρουσία στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης των κρατών μελών ε, μάλλον ο κανονισμός λέει ότι ε, δεν μπορούν να είναι κάτω από δύο και όχι πάνω από 18. Ίσως το 18 να είναι το όριο για την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάντως παραμένει ανοιχτό ένα πρόβλημα που πρέπει να δούμε και έχει υπογραμμιστεί πολλές φορές των σχέσεων μεταξύ των δύο δικαστηρίων επ' αυτού πρέπει να, να περιμένουμε λίγο αλλά και της ευρωπαϊκής ψυχής. Εμείς λέμε στο άρθρο 2 της συνθήκης ότι στηριζόμαστε στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ε, να σκεφτούμε λοιπόν και την έννοια αυτή του ανθρώπου, τα όρια της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, των ορίων του. Πέραν αυτού, συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενο της ε, εκθέσεως. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει κυρία Κοπά για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή ένωση είναι και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου και του ρόλου του στην προάσπιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ελπίδα όλων μας είναι η διάσκεψη της Καμπάλα που θα αναθεωρήσει το καταστατικό της ρώμης να αποτελέσει πραγματικό σταθμό για την περαιτέρω εξέλιξη του δικαστηρίου. η διεθνή κοινότητα καλείται να ενισχύσει το κύρος του θεσμού και να εξασφαλίσει την προστασία και περαιτέρω ενίσχυση τη ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα τη διεθνού ποινική δικαιοσύνη στα πλαίσια της αναθεωρητικής διαδικασίας έχουν ήδη παρουσιαστεί διάφορες προτάσεις με αναμφισβήτητα πιο σημαντική αυτή που αφορά το έγκλημα της επίθεσης. αυτό που προέχει σήμερα ωστόσο είναι να γίνει σαφές ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο επιθυμεί να τονίσει πως τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν μπορούν να παραμένουν ατιμόρυτα αυτό που θέλουμε είναι σαφήνεια δικαίου και συνεργασία από όσο το δυνατο περισσότερα κράτη μέλη της διεθνούς κοινότητας ώστε να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία μέσα από μια δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία. οι εγκληματίες πολέμου πρέπει να είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. είναι αυτή η βεβαιότητα της ποινής που μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή παρόμοιων πράξεων στο μέλλον αλλά και να ανοίξει το δρόμο για τη συμφιλίωση μετά από βίαιες συγκρούσεις επιβεβαιώνουμε λοιπόν την απόλυτη στήριξή μας στους σκοπούς του δικαστηρίου και την προσήλωσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ευχόμενοι κάθε επιτυχία στην αναθεωρητική διάσκεψη της ουγκάντα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κατσμάρεκ για 1,5 λεπτό. Pani Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά την διεθνή συνδιάσκεψη και την δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προστασία των αξιών μας, πιστεύω ότι οι εγκληματίες, αυτοί που διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σαφώς και θα πρέπει να προσαχθούν σε αυτό το ποινικό δικαστήριο το οποίο δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό. Άτομα όπως ο Σαντάμ αλλά και άτομα που σήμερα συνεχίζουν να είναι ελεύθερα ενώ έχουν διαπράξει εγκλήματα στο Σουδάν και αλλού στην Αφρική θα πρέπει να προσαχθούν και βεβαίως αν είχαμε ένα τέτοιο δικαστήριο πριν από 70 χρόνια ίσως και η δολοφονίες στο κάτι να είχαν αποφευχθεί. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα πρέπει να ενισχυθεί και όλοι αυτοί οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας να τιμωρούνται. Και βεβαίως και θα πρέπει το καθεστώς αυτής της συνθήκης μέσω της αναθεώρησης που θα γίνει στην Ουγκάντα να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκόμες. Για ένα λεπτό. Η κυρία Γκόμες. Η, η σύνοδος της Καμπάλα παίζει ένα σημαντικό έχει σημαντικό ρόλο για την αλλαγή ε, του καταστατικού του Διεθνούς Δικαστήριου. Όταν όμως μιλάμε για την απαγγελία κατηγοριών κατά του Μπασίρ, μπαίνουν και άλλες διαστάσεις στη συζήτηση. Έχουν τονιστεί, έχει τονιστεί το ότι ο, ή έχει υπογραμμιστεί το ότι έχει, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κατά του πρόεδρου του, Σουδάν. Οι παρατηρητές των Σουδανικών εκλογών είπαν ότι ο τρόπος εξαγωγής τους δεν ήταν διεθνώς αποδεκτός, αποδεκτή. Ε, δεν τηρούσαν τα διεθνή στάνταρ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σαφής επίκληση της δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αντιφάσεις. Ο Αλμπασίρ πρέπει να δικαστεί. Και αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα για να εμποδιστούν άλλοι δικτάτορες από τη... το να πλήττουν το δικό τους λαούς. Δυστυχώς κάτι τέτοιο, αλλιώς κάτι τέτοιο θα έχει αρνητικές συνέπειες. Το λόγο έχει ο κύριος Μαρκοβέη για 1,5 λεπτό. Η κυρία Μαρκοβέη. Ευχαριστώ. Θα, μιλήσω για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και θα ήθελα να σας μιλήσω και με την ιδιότητά μου του νομικού. Να ευχαριστήσω την προσοχή σας στο ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και μάλιστα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή αυτή σύμβαση, ε, υπάρχει απέτηση ο ετών να εξαντλήσει τα εγχώρια ένδικα μέσα πριν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα θα πρέπει το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση να έχει την ευκαιρία να αποφανθεί ως ε, τελευταία αρμόδια, αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο προτού πάει το θέμα στο δικαστήριο του, του Στρασβούργου. Και θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να ε, τηρήσουν όλα αυτά τα προαπαιτούμενα. Θα πρέπει δηλαδή το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου να έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τη σύμβαση σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην ξεχνάμε ότι έτσι έχει εφαρμόσει τη σύμβαση αυτή το Δικαστήριο ε, όλα αυτά τα χρόνια. Να σας υπενθυμίσω επίσης τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, στην περίπτωση ε, των ευρημάτων στο Βόσπορο σε σχέση και με την αεροπορική εταιρεία και το θέμα της Ιρλανδίας. Ό,τι δηλαδή είναι ισότιμο. Ισότιμο είναι η λέξη κλειδί στην απόφαση του δικαστηρίου. Θα ήθελα λοιπόν να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά τη διαδικασία που ε, θεσμοθετούμε αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να λειτουργήσουμε προς το συμφέρον των πολιτών αλλά και να διατηρήσουμε τα καλώς κείμενα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ε, Ράντζελ. Ενάμιση λεπτό μάλλον. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, ικανοποίηση ε, που νιώθουν οι Πορτογάλοι βουλευτές του ΕΛΚ, διότι έχει πλέον ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της προσχώρησης ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, ΕΣΤΑ, στη σύμβαση αυτή. Μία χώρα σαν την Πορτογαλία ανέκαθεν έχει υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ νωρίς καταργήθηκε η δουλεία στην Πορτογαλία, πολύ νωρίς καταργήθηκε η θανατική ποινή στη χώρα μου. Ανέκαθεν λοιπόν η χώρα μου ήταν υπερασπιστή της ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα κάνει το παν ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο λοιπόν να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΤΑ. Από νομικής, πολιτικής, ε, συνταματικής πλευράς όλο αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επομένως θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσδίδουν στο όλο θέμα τη σημασία που του αξίζει. Πρέπει να αποστείλουμε σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και να δείξουμε στα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο ε, ισχυρή είναι η φωνή μας και πόσο θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξεκινάμε λοιπόν με το Catch the Eye, SPARP, ε, για ένα λεπτό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες ε, δεν περιλαμβάνονται πλέον ε, περιλαμβάνονται και γίνονται σεβαστά από όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα βήμα προς τα εμπρός ε, αφορά τις ελευθερίες όλων των πολιτών, προσφέρει τη θέμενη αξία και ο στόχος μας πρέπει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου τα, οι προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί το βασίλειο της ελευθερίας. Το αντίθετο θα αποτελούσε παραβιάσεις σημαντικών ελευθεριών. Και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να λαμβάνει η χώρα συστηματικά. Πρέπει λοιπόν να συστήσουμε τις ε, κατάλληλες διαδικασίες ε, για τα ε, δικαστήρια και το δρόμο που πρέπει να ακολουθούν. Το ρόλο έχει ο κύριος Ζέμκε για ένα λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά που συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι η Αφρική είναι μια ήπειρος όπου πολύ συχνά γίνονται ε, δολοφονίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς λοιπόν το ε, Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην ε, περίπτωση αυτών των εγκλημάτων, τα οποία δεν μπορούν να παραμένουν ατιμόρυτα. Εγώ λοιπόν είμαι ένας από εκείνους οι οποίοι κατηγορηματικά υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οφείλουμε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε ε, να καταστεί ε, ακόμα πιο αποτελεσματικό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Φλάσιο Μπενκόβα, Γιώβα. Κυρία Υπουργέ, όπως ε, ήδη αναφέρθηκε, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, σύμβαση αυτή είναι συμβολική γιατί πιστεύω ότι θα ενισχυθεί η ουσία αυτής της σύμβασης και εκτός αυτού θα υπάρχει και μια πρακτική σημασία στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταργηθούν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν υποχρεωμένη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικό όχι μόνο να προστατεύσουμε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι υπόκεινται στην ευρωπαϊκή νομολογία. Είμαι λοιπόν ευτυχής για το ότι ε, πρέπει να τηρούνται όλες οι ρήτρε της ε, σύμβασης αυτής. Και αυτό που έχει σημασία είναι να επισημανθούν τα προβλήματα που συνεπάγεται όλη αυτή η διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, μη κρατική οντότητα δεν πρέπει να ζητήσει περιττές τροποποιήσεις. Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο είναι ήδη επιβαρημένο, γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να αποφύγουμε τη διάπραξη λαθών. Ευχαριστούμε πολύ. Μορβάη, ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, είμαι νέο κοπομέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αρχίζω να συνηθίζω σιγά σιγά. Δηλαδή στο ότι ε, κάθε συζήτηση ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Συνήθως εδώ στις συζητήσεις δεν παρίστανται πάνω από 20 έως 30 άτομα παρότι είμαστε 700 τόσοι Ορισμένοι από εμά δεν ακολουθούν την κομματική γραμμή κατά τις ψηφοφορίες αλλά ακολουθούν αυτά που μας ε, επιβάλλει η συνείδησή μας. Και όταν υποβάλλουμε ερωτήσεις στην Κομισιόν, συνήθως δεν παίρνουμε ερωτήσεις. Και απευθύνομαι σε εσά, κύριε Επίτροπε. Είσαστε αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ να ε, κάνετε μία εξαίρεση αυτή τη φορά και να μου δώσετε μία συγκεκριμένη απάντηση. Και η ερώτησή μου είναι η εξή. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία ε, στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί συνυπογράφει την ε, ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη στιγμή που την έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη. Πετε μου, τι θα προκύψει, ποιο όφελο θα προκύψει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα υπάρξουν κάποιε εξελίξει. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ λοιπόν να ε, κάνετε μια εξαίρεση στον κανόνα και να μου δώσετε μια τίμια απάντηση. Ματέρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Επίτροπε προσχώρηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημαίνει ότι θα έχουμε μία ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών τόσο μέσα στο εσωτερικό των 27 κρατών μελών όσο και στο εξωτερικό. Αν σκεφτούμε όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε αυτή την ευκαιρία την οποία εμείς περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Η νομολογία τόσο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσο και του Δικαστηρίου του Στρασβουργού εδώ και καιρό ε, έχουν βάλει, έχουν θέσει τις βάσεις ε, για αυτή την ε, μετάβαση, μια πραγματική μετάβαση για όλους μας. Θέλω να αναφερθώ στην σημασία που θα έχει αυτή η πράξη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι θα μπορούν να καταφύγουν ε, στο ε, δικαστήριο του Στρασβούργου και θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη προστασία. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι η αυτονομία των δύο αυτών δικαστηρίων πρέπει να παραμείνει ανέπαφη και θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον εισηγητή για την έκθεσή του. Επίσης ε, να αναφέρω ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους διαθεσμούς όπου βέβαια ο κάθε ένας από αυτούς θα σέβεται τις αρμοδιότητες του άλλου. Ευχαριστούμε. Ε, κύριος ε, Ντεβίγκο έχει ζητήσει το λόγο. Δύο διευκρινήσεις. Καταρχάς, τα άρθρα της χάρτας που είναι ίδια με τα αντίστοιχα άρθρα της σύμβασης, σύμβασης είναι τα ίδια και σημαίνουν το ίδιο πράγμα. 52 και 53. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ίδιες λέξεις, ίδιο νόημα. Επίσης είναι υπερεθνική η δικαιοδοσία στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Πρέπει να πάει στο δικαστήριο κανείς του Στρασβούργου με την προδικαστική διαδικασία. Ε, εν πάση πτώση διαβάστε την έκθεση του κυρίου Χαουρεγκή διότι είναι σαφή τα πράγματα. Εάν θέλετε να κατακρίνετε, κατακρίνετε, αλλά διαβάστε πρώτα την έκθεση. Έκλεισε η συζήτηση. Κατόπιν τούτου θα θέλω να δώσω στον κύριο Λόπε Καρίντο, ε, εξ ονόματος ε, του Συμβουλίου, υφυπουργό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναφορικά με το πρώτο σημείο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θα ήθελα καταρχάς να επαναλάβω τα συγχαρητήριά μας στους εισηγητές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τόσο γρήγορα δούλεψαν και παρουσίασαν αυτό το σχέδιο εντολής για τη διαπραγμάτευση. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Άντριου Νταφ, ο οποίος είπε σαφέστατα ότι η καινούργια κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ακολουθεί κατά γράμμα τη γραμμή αυτή και συμφωνεί να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΣΤΑ εφαρμόζοντας και τα περιεχόμενα της ειδικής της Λισαβόνας. Ωστόσο, άλλοι συμπατριώτες του κυρίου Νταφ δήλωσαν το αντίθετο. Εκπρόσωποι της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, αλλά και ο εκπρόσωπος της ομάδας Ευρώπη για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ο εκπρόσωπος του τελευταίου βεβαίως δεν είναι Βρετανός πολίτης. Έχουμε και την κυρία Σιγκλέρ αλλά και την κυρία Μορβάη, οι οποίες ρώτησαν σαφέστατα γιατί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει και να επικυρώσει αυτή τη σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη είναι μέρη, είναι μέλη της σύμβασης αυτής. Η απάντηση είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ασκούν αυτή την εξουσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί αυτή την εξουσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει αρμοδιότητα, έχει εξουσία την οποία τις έχουν εκχωρήσει τα κράτη-μέλη. Δεν αρκεί λοιπόν τα κράτη-μέλη να ε, υπογράψουν τη σύμβαση αυτή. Χρειάζεται ε, να την υπογράψει τη σύμβαση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό πρόσωπο. Ακριβώς για να ε, επικρατήσει η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια και να ε, χαίρει πλήρους προστασίας η νομική αυτή έννοια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αρνούνται ε, την ύπαρξη υπερεθνικού ελέγχου πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τελείως αντιφατικό αυτό. Εάν κάποιος νομίζει ότι ε, ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κακό ή ότι υπάρχουν διάφοροι πολύ κακοί γραφειοκράτες οι οποίοι ε, λειτουργούν με πολύ άσχημο τρόπο τότε πώς είναι το ίδιος άνθρωπος να αρνείται τον έλεγχο, τον υπερεθνικό έλεγχο ε, σε αυτά τα όργανα ή σε αυτά τα στελέχη ή σε αυτό το μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ε, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Και πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα να υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μεντελεβίβο. Πράγματι η Επιτροπή λειτουργήσε πολύ γρήγορα, το Συμβούλιο λειτουργήσε γρήγορα και σίγουρα θα εγκριθεί η εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων στις 4 ε, ε, Ιουνίου στην, ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Τώρα, Πολύ σημαντικό είναι το θέμα του Διεθνούς Δικαστηρίου στη διάσκεψη για την αναθεώρηση και μιλώ εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου η οποία θα είναι παρούσα, θα εκπροσωπηθεί σε αυτό το φόρουμ και θα υπογραμμίσει σαφέστατα ότι τα κράτη-μέλη πρέπει, οφείλουν να συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση συμφωνούμε με έναν από τους βασικούς στόχους της διάσκεψης αυτής. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι το ότι δεν θα μπορεί πλέον να καθυστερεί κατά 7 χρόνια η έκδοση ε, ε, διαφόρων κατηγορημένων για εγκλήματα πολέμου. Επίσης ε, θα μπορούσε η εμπορία όπλων σε περιπτώσεις σύραξης και συγκρούσεων να θεωρείται αυτή καθεαυτή ως έγκλημα ε, πολέμου. Θα έχουμε λοιπόν ως στόχο την, ε, τον ορισμό του αδικήματος της επίθεσης. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι παρόν στη διάσκεψη της Καμπάλα θα είναι παρόν σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα πολιτική σημασία, έχει μεγάλη συμβολική σημασία αλλά και νομική σημασία γιατί θα ληφθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη διατύπωση νομικών κειμένων. Είναι πολύ καλό που έγινε αυτή η συζήτηση σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε και να ε, επαναλάβουμε τις βασικές αρχές που μας ενώνουν όλους. Άλλωστε γνωρίζουμε όλοι πόσοι ε, έχουν υποφέρει και πόσο σημαντική είναι η αλλαγή του καταστατικού της Ρώμης ώστε πλέον να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η Επίτροπος η κυρία Ρέντινγκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Χάρτα Βασικών Δικαιωμάτων και η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι θαυμάσια κείμενα. Αποτελούν τη βάση των αξιών πάνω στις οποίες εμείς οικοδομήσαμε την κοινωνία μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ιστορικά και γι' αυτό δεν θα πρέπει που δεν είναι να οδηγήσουν σε μια κομματική πολεμική. Και ομολογώ ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη πραγματικά που αυτή τη στιγμή της οικοδόμησης Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να προχωρήσουμε θέτοντας σε ισχύ την Χάρτα των Βασικών Δικαιωμάτων και εντασσόμενη στην Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ακούγοντας τι έχει να πει ο κύριος Λόπες Καρίχο, ο εισηγητής και οι συνεισηγητές και η και Καρίδα έχουν πει εδώ στο Κοινοβούλιο, κατανοώ ότι και εσείς έχετε πλήρη επίγνωση του ιστορικού έργου που έχουμε πια στα χέρια μας. Η προστιθέμενη αξία της ένταξης εξηγήθηκε σαφέστατα και στα εν και στις συμβολές πολλών εκ των βουλευτών. Τα κράτη-μέλη έχουν όλοι προσυπογράψει την σύμβαση αλλά επίσης όπως εξήγησε ο κ. Υπουργό μόλις τώρα, έχουν μεταφέρει σημαντικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είναι φυσιολογικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δρά ως Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάγεται στους ίδιους ελέγχους των ειδικών δικαστηρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως και τα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Ενδεχομένω θα μπορούσε να υπάρχει μια απόφαση Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά μια βιομηχανία στον τομέα του ανταγωνισμού που θα μπορούσε ενδεχομένω άμεσα να γίνει προσφύγη κατά στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Αυτό σήμερα δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να γίνει. Και υπάρχουν πολλά άλλα συγκεκριμένα παραδείγματα που τονίσατε. Συγκεκριμένα παραδείγματα που θα βοηθήσουν τους πολίτες. Γιατί, και αυτό είναι κάτι καινούριο, γιατί λέω θα έχουν μια διπλή εγγύηση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου που θα κρίνει βάσει της χάρτας βασικών δικαιωμάτων που είναι παρεμπιπτόντως δεσμευτικό για όλα τα κρατη πρέπει να πούμε αυτό ξεκάθαρα και δεν μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος ο οποίος ε, έχει εκλεγεί από πολίτες και έχει μια εντολή εκλεγμένου μπορεί να διαμφισβητεί τα δικαιώματα αυτών των πολιτών. Είναι καλύτερα να έχουν δύο φορές τα δικαιώματά τους οι πολίτες παρά να μην τα έχουν καμία φορά. Εδώ τους δίνουμε δύο φορές το δικαίωμα και αυτό σημαίνει Ευρώπη. Η Ευρώπη σημαίνει δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και χαίρομαι που το σώμα προασπίζει αυτά τα δικαιώματα. Ναι, θα έχουμε τώρα μια χάρτα βασικών δικαιωμάτων όπου οι πολίτες θα ξέρουν ότι μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια για να μπορούν τα δικαιώματά τους να ληφθούν σοβαρά υπόψη. το θέμα κατά πόσον τώρα θα πρέπει, δεν θα πρέπει να είμαστε τμήμα της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι πια ερώτημα γιατί το άρθρο 6 της συνθήκης υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενταχθεί στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται πια να το συζητάμε. και θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι αυτή η ένταξη θα αφήσει ως έχει την θέση των κρατών μελών έναντι της σύμβασης δεν θα αλλάξει τίποτα εφόσον δεν διακυβεύεται καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό αφορά λοιπόν τις σχέσεις κράτους και σύμβασεις που δεν θα αλλάξουν, θα υπάρχουν μόνο τώρα συμπληρωματικές εγγυήσεις όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο. Το θέμα της, ε, των συγκρουμένων ε, δικαστικών συστημάτων θα πρέπει να αναλυθεί και ευχαριστώ τον εισηγητή που το εξέτασε. Μέχρι στιγμής είδαμε ότι αυτές οι συγκρούσεις είναι ελάχιστες. Γιατί η σύμβαση ήδη είναι τμήμα των νόμων που λαμβάνει υπόψη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και η σύμβαση θα λειτουργήσει σαν ένα ελάχιστο πρότυπο και η Εκτελεστική Επιτροπή αναμένει ότι τα δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου θα ε, συγκλίνουν τις απόψεις τους προσεχώς. Όσον αφορά τα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα, Πρόεδρε, βέβαια, όσον αφορά τα θέματα δικαστική διαμάση, δεν είναι θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή του συστήματος του δικαστηρίου συγγνώμη στην, στο Λουξεμβούργο είναι θέμα του Βρετανικού συστήματος και τους έχουμε ζητήσει να αναθεωρήσουν το θέμα όπου πολλές φορές, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, μπορεί να είναι πάρα πολύ νοητικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τη στιγμή, υπό την των εισηγητών του, εργάστηκε πάρα πολύ θετικά και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συνοδεύει μια διαδικασία η οποία οπωσδήποτε θα είναι δύσκολη, θα είναι χρονοβόρα όπου θα πρέπει να επιληθούν τεχνικά προβλήματα και ξέρετε ότι τεχνικά προβλήματα μπορούν να καταστούν και πολύ πολιτικά. Εγώ βασίζομαι λοιπόν στο Κοινοβούλιο να συνεχίσει να μας συνοδεύει σε αυτό το τόσο δύσκολο έργο. Και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, το, και, την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα το αφήσω στα δικά σας χέρια. Αν χρειάζεται χέρα βοηθείας θα είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά αυτό είναι θέμα της αυτονομίας των βουλευτών να βρουν ένα κοινό έδαφος με τους συναδέλφους και δεν θα πρέπει να είναι και τόσο δύσκολο φαντάζομαι. Πρόεδρε, όσον αφορά την ICC, το Κοινοβούλιο υποδέχθηκε τον εισαγγελέο Κόντορ και τον πρόεδρο του δικαστηρίου κ. και νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της Ευρώπης. Και πιστεύουμε ότι η διάσκεψη της Καμπάλα είναι η πιο σημαντική διεθνής διάσκεψη για το διεθνές δίκαιο εδώ και δεκαετίας και θα πρέπει λοιπόν να της αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία και βασίζομαι και εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί ξέρω ότι θα είναι παρόντες ευρωβουλευτές και θα πάρουν και το λόγο στην Καμπάλα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε και θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σωματώνοντας τα αποτελέσματα της διάσκεψης στις ε, πολιτικές του για τη διεθνή δικαιοσύνη, στην, για την ενίσχυση προς τρίτες χώρες και κυρίως για όλες τις διαπραγματεύσει που θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Ιδίως θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την δημιουργία εθνικού δυναμικού για να ενδυναμώσουμε τα εθνικά δικαστικά συστήματα να μπορούν να πραγματοποιούν τις απαραίτητες έρευνες. Η δική μας πολιτική στον τομέα αυτό δεν αλλάζει, ούτε μειώνεται. Αλλά έχουμε ένα νέο μέσο στη διάθεσή μας και αυτό το νέο μέσο είναι η συνθήκη της Λισαβόνας που μας δίνει νέες δυνατότητες να είμαστε πιο συνεπείς και πιο αποτελεσματικοί στην υποστήριξή μας των δικαστηρίων και ευθυγρασμένη με την ενθάρρυνση του Κοινοβουλίου όπως εκφράζεται στο ψήφισμα και όπως εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτηση είπατε εκπρόσωπος αντιπρόεδρος και οι υπηρεσίε της θα συνεχίσουν να προωθούν αποτελεσματικά την ε, γενική ε, πρόσβαση στο καταστατικό της Ρώμης. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό με τους εταίρους μας εκτός της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, υπήρχαν δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα μου επιτρέψετε σύντομα να απαντήσω. Η πρώτη ήταν κατά πόσον ένα ένταγμα σύλληψη κατά του Πρόεδρου Αλμπασίρ είναι τμήμα της λύσης ή τμήμα του προβλήματος. Η Κομισιόν προφανώς θεωρεί ότι αυτό είναι ένα τμήμα μιας μακροπρόθεσμης λύσης, γιατί το αυτό αυτοσύλληψης καταδεικνύει ότι με την έδρυση του δικαστηρίου είναι άμεση η δικαιοσύνη. Άσχετα το για ποιον πρόκειται, ακόμα και αν το άτομο αυτό είναι επικεφαλής ενός κράτους. Και ακόμα και αν αυτό το ένταλμα σύλληψης δεν ε, εφαρμοστεί αμέσως, δεν θα εξαφανιστεί, γιατί η Ρόησης είναι ένα μόνιμο δικαστήριο και θα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να καλεί το Σουδάν να συνεργαστεί απόλυτα με το δικαστήριο. Το θέμα του κατά πόσον η Εκτελεστική Επιτροπή θα υποβάλει τροπολογίες σε συνάντηση Καμπάλα ε, μπορεί να απαντηθεί με όχι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέρος, τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που θα διαπραγματευτούν τις τροπολογίες Παρ' όλα αυτά η Εκτελεστική Επιτροπή θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην καταγραφή των αποτελεσμάτων της διάσκεψης και βασιζόμαστε απόλυτα στην Ισπανική Προεδρία για να ηγηθεί των ευρωπαϊκών κρατών ούτω ώστε η φωνή τους να εισακουστεί και να είναι πολύ αποτελεσματική στα πλαίσια της διάσκεψης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Την Επίτροπο εισηγητής για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρεμβαίνοντες, διότι οι περισσότεροι εκδήλωσαν τη θετική τους στάση ως προς την ε, Συμφωνία Προσχώρησης, την οποία θα ψηφίσουμε αύριο. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επίτροπο, την κυρία Ρέντιν, για την ευκαιρία που είχαμε να δουλέψουμε και να συνεργαστούμε είναι περίπλοκη η διαπραγμάτευση και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την παρακολουθήσει στενά. Ε, συντομία, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιε διευκρινήσει. Η προσχώρηση δεν είναι μόνο συμβολική σημασία. Έχει νομική σημασία, νομική αξία. Ε, ποια είναι η προστιθέμενή τη αξία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γίνεται διαγωνισμός για μόνιμους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ας πούμε ότι γίνεται διάκριση εις βάρος νομικών, είτε για τεχνικούς λόγους, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Πού μπορούν να προσφύγουν οι άνθρωποι αυτοί. Στο δικαστήριο. Τι, τι προσθέτει η προσχώρηση αυτή. Ότι το δικαίωμά τους στην ισότητα δεν αναγνωρίστηκε. Είναι ένα νέο δικαστήριο και μια νέα ευκαιρία για να εγγυηθούμε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι ε, το θέμα της ισότητας. Δεν είναι δηλαδή συμβολική μόνο η συνεισφορά της προσχώρησης στη σύμβαση αυτή, είναι και ουσιαστική, έχει νομική αξία. Τα μέλη του Κοινοβουλίου είπαν ότι επιθυμούν η διαπραγμάτευση να μην ε, στραφεί μόνο ως προς, ε, στο θέμα της προσχώρησης στη σύμβαση αλλά να ασχοληθεί και με τα πρωτόκολλα τα οποία έχει ενσωματώσει με την πάροδο του χρόνου η σύμβαση αυτή και μιλούμε επίσης και για τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο τα δύο έγγραφα, η σύμβαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, θα, ε, θα θεωρούνται ότι έχουν ισότιμη αξία. Και μιλούμε για μια αμοιβαία αναγνώριση του οικομενικού συστήματος προστασίας ε, των δικαιωμάτων του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένης και της χάρτας του Τωρίνο. Ευχαριστώ.